Σας παρακαλώ εγώ ίδιος προσωπικά και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πόσο σημαντική είναι αυτή η συγκυρία. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Και τώρα προχωρούμε στην ημερησία διάταξη. Έχουμε το τελικό σχέδιο με τις διατάξεις που 22 Σεπτεμβρίου είναι κρίθη σύμφωνα με τη διάταξη 137. Δεν έχουμε ενστάσεις, παρατηρήσεις, επιφυλάξεις για τροποποίηση σε σχέση με αυτό το τελικό σχέδιο της μερική διατάξεως. Όχι, επομένω. θεωρώ ότι η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Οπότε και τώρα προχωρούμε παρακάτω.